ρόλο. Ο κ. Ρέγγλ μας έδινε διδάγματα και μαθήματα σε, ό, όλους, σε όλους και για όλα, αλλά ποτέ δεν ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, στην ε, πραγματικότητα δηλαδή ήταν στο περιθώριο οποιοδήποτε κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η εμπειρία της λειτουργίας τα τελευταία χρόνια ήταν από τις πιο αρνητικές. Ε, το είδαμε ότι ε, η, τα μνημόνια έγιναν εις βάρος πολλών πολιτών και με τρόπο πάρα πολύ ακριβό. Ε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια σε βάθος μεταρρύθμιση του μηχανισμού. Εμείς είχαμε προτείνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να συνεισφέρει στους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να ασκούμε δημοσιονομικό έλεγχο στις δραστηριότητές του. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Παρ' όλα αυτά έχουμε υποβάλει τροπολογία και θα ψηφιστεί. Δεύτερο, δεύτερη πρότασή μας για το κείμενο ε, ήταν στα μελλοντικά προγράμματα ε, να, ε, τα μελλοντικά προγράμματα να είναι μέσω, να εγκριθούν μέσω κατεξιότηση πράξεων. και αυτό για να έχουμε περισσότερο έλεγχο. Ούτε αυτό εγκρίθηκε και έχουμε υποβάλει τροπολογία. Άλλη τροπολογία που βάλουμε είναι να γίνει μια ανάλυση κοινωνικού αντικτύπου στη, της πολιτικής και των πράξεων του μηχανισμού. Δεν έγινε στην Ελλάδα και γι' αυτό είδαμε τι καταστροφή επικράτησε. Επίσης χρειαζόμαστε περισσότερο έλεγχο στο διορισμό του διευθυντή. Θέλουμε μια διαδικασία πραγματικά δημοκρατική και να έχουμε διάφορες επιλογές. Τέλος, το θέμα του backstop. Ένα backstop θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο ε, δεν θα λειτουργήσει αν, αν απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Θέλουμε το backstop να γίνεται αυτομάτως με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ένα backstop το οποίο υπόκειται στην ομοφωνία του Συμβουλίου δεν θα λειτουργήσει. Οπότε δεν είμαστε ικανοποιημένοι ούτε με την μεταρρύθμιση ούτε με την έκθεση. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ο κ. Παπαδημούλης. Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό ταμείο σταθερότητας. ναι το χρειαζόμαστε και γι' αυτό ακριβώς δεν χρειαζόμαστε κύριε ντομπρόφσκης ένα ευρωπαϊκό αντίγραφο μια ευρωπαϊκή ρεπλίκα του διεθνούς νομισματικού ταμείου. και σας το λέω εγώ γιατί στην ελλάδα ζήσαμε οδυνηρά στην πλάτη του ελληνικού λαού τις οδυνηρές συνέπειες από τις λάθος νεοφιλελεύθερες συνταγές και τους λάθος πολλαπλασιαστές του διεθνούς νομισματικού ταμείου. και χρειαζόμαστε τώρα ένα ευρωπαϊκό ταμείο σταθερότητας που όπως είπε και η κυρία χούμπνερ πρέπει να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή ένωμη τάξη να δουλεύει με την κοινοτική μέθοδο και να λογοδοτεί και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και όχι απλώς στα εθνικά κοινοβούλια και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο γιατί αυτό δεν εξασφαλίζεται με την μέθοδο την διακυβερνητική αλλά την κοινοτική και επιπλέον πρέπει όχι απλώς να αντικαταστήσει το διεθνές νομισματικό ταμείο αλλά να αντικαταστήσει και τη συνταγή του διεθνούς νομισματικού ταμείου το δόγμα σόιμπλε τον νεοφιλελευθερισμό. και γι' αυτό χρειαζόμαστε να τρέξουμε και θετικές αλλαγές για να λογοδοτεί όχι μόνο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αλλά και στο ελεγκτικό συνέδριο και χρειαζόμαστε και έναν αντιπρόεδρο της κομισιόν αρμόδιο για τα θέματα της ευρωζώνης όχι μόνο της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής. αν δεν τα κάνουμε αυτά θα είμαστε πολύ πίσω από τις απαιτήσει. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Παπαδημούλη, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βάλη εξ ονόματος του EFDD. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορούμε ως πολιτική ομάδα να αποδεχθούμε τη βάση της λογικής του σκεπτικού για τη θέσπιση αυτού του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Και αυτό διότι πρόκειται για ένα απλό αντίγραφο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα που απλώ επισημοποιείται τώρα εδώ πέρα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Και προβλέπεται εδώ πέρα ότι υπό προποθέσει θα δίνει δάνεια. Κύριε Παπαδημούλε, μην ξεχνάμε όμω ότι τα δάνεια αυτά ακριβώ ταπείνωσαν τον ευρωπαϊκό λαό τα χρήματα αυτά τα οποία δόθηκαν προς την ε, Ελλάδα προκειμένου να γίνουν μεταρρυθμίσεις με ιδιαίτερο πόνο, οδύνη, με αίμα και υδρότα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν πώς λειτουργήσαν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί στο παρελθόν. Και τώρα θέλουμε να τους επισημοποιήσουμε κάνοντας τους δήθεν πιο δημοκρατικούς δεν συμφωνούμε με αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλη αυτή τη δομή και να δούμε πραγματικά ποιε είναι οι πραγματικέ ανισορροπίε στο πλαίσιο τη Ευρωζώνη. Άλλα μέσα χρειαζόμαστε. Μια πραγματική δημοκρατία. Αλλά δυστυχώ δεν απορρέει κάτι τέτοιο από τη θέσπιση αυτού του νέου οργάνου. Ευχαριστώ. E Ο Μίχαλ Μαρούσικ, εξ του ΕΝΕΦ, e για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γίνεται λόγος για την ενιαία αγορά αυτή τη στιγμή και η βάση της ενιαίας αγοράς είναι το να μπορούμε να έχουμε συστήματα τα οποία λειτουργούν σωστά και που δεν χρεοκοπούν. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι απουσιάζουν οι μηχανισμοί αυτοί οι οποίοι θα επιτρέψουν να έχουμε επικερδείς ανθούσες αγορέ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε παραγικότητα χαμηλού κόστου και να μπορούμε να αποκρινόμαστε στι ανάγκε των καταναλωτών. Οι δύο αυτέ αρχέ αρκούν από μόνες του. Όποιεδήποτε άλλε παρεμβάσει στην αγορά κάνουν κάποιε ανεπαρκεί και ανίκανε τελικά επιχειρήσει απλώ να επιβιώνουν. Ενώ ζημιώνται τελικά με περισσότερους φόρους και κόστος οι υγιείς επιχειρήσεις. Ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα είναι ένας ακόμα οργανισμός ο οποίος θα παρεμβαίνει τεχνητά στην ελεύθερη λειτουργία της ενίας αγοράς. Και το αποτέλεσμα θα είναι ένα και μοναδικό. Στην πράξη θα έχουμε Επιχειρήσει οι οποίες δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν σωστά, οι υγιείς επιχειρήσεις δεν θα ανθούν οικονομικά, ενώ αυτές που θα έπρεπε να χροκοπήσουν απλώς θα επιβιώνουν με τρόπο εντελώ τεχνητό. Το να δώσουμε περισσότερα κονδύλια σε έναν τέτοιο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ουσιαστικά θα προωθήσει τη δράση συγκεκριμένων ολιγαρχών μέσω συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε τέτοιους μηχανισμούς οι οποίοι θα τιμωρήσουν ουσιαστικά τι υγιεί επιχειρήσει και θα επιβραβεύσουν τη μη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρούσικ. Ε, από την ομάδα των μη εγγεγραμμένων, κυρία Σοφή Μοντέλ. Συνάλφη, το 2010 η Τρόικα, η Κομισιόν δηλαδή, η Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επέβαλε αυστηρο... δημοσιονομική αυστηρότητα στον ελληνικό λαό και τον έριξε στην ε, μιζέρια. Αυτό το... Αυτή η εικόνα προφανώς σας άνοιξε την όρεξη και θέλετε περισσότερο από τα ίδια. Ε, η αποστολή αυτού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα ε, λέγεται ότι είναι η βοήθεια, ε, χρηματοπιστωτική βοήθεια στα κράτη-μέλη που το χρειάζονται και υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Σύμφωνα με το πρόγραμμα διάσωση. Τα προγράμματα διάσωση όμω ξέρετε τι σημαίνουν. Στην Ελλάδα μειώθηκαν πάρα πολλοί συντάξει, οι μισθοί το ίδιο, ιδιωτικοποιήθηκαν οι, οι δημόσιε εταιρείε και βέβαια ε, εκτινάχθηκε η ανεργία. Ε, η, και όλα αυτά υπό τις διαταγές της ε, Γερμανίας. Μία, ένα είναι σίγουρο. Ε, δεν χρειάζεται αντίδραση στη Γαλλία, αρκείτε εσείς για να καταστήσετε την Ευρώπη ακόμα πιο δυσάρεστη στους πολίτες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μόντελ. Αυτή ήταν εκπρόσωποι των ομάδων. Τώρα περνάμε στις ομιλίες των συναδέλφων. Και ο πρώτος είναι ο κύριος Φέρμερ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Κατά την κρίση του δημοσίου χρέους και του οικονομικού συστήματος διαπιστώσαμε ότι ο Ευρωπαϊκός ε, Μηχανισμός Σταθεροποίησης και ο προκάτοχος του EFSF απέδειξαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν με μη πολιτικοποιημένο τρόπο και με βάση στοιχεία και με βάση σαφείς κανόνες ε, είχαν αποτέλεσμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το τονίσουμε ότι είναι η βάση και των νέων προτάσεων της Κομισιόν. Ο EFSF και ο ESM επέτυχαν σε όλες τις χώρες που είχαν πρόβλημα. Οπότε, ε, λογικό πόρισμα, αυτό το οποίο λειτουργεί δεν θα πρέπει να αμφισβητείται. Μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα είναι οι σχέσεις ε, μεταξύ ε, ενό τέτοιου μηχανισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, μέσω μια διοργανική συμφωνία. Αλλά μην τα παρακάνουμε. Διότι σε τελευταία ανάλυση πιστώσει δίδονται από τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλο τα... οι εθνικοί προπολογισμοί και τα εθνικά κοινοβούλια είναι εκείνοι οι οποίοι ε, από τη μία δίδουν τους πόρου και από την άλλη πρέπει να ελέγχουν. Αυτή είναι η αρχή τη ε, Ευθύνη. Και ορισμένε προτάσει των συναδέλφων ότι θα έπρεπε με πλειοψηφία να αποφασίζουμε για προγράμματα μακροοικονομικής ε, προσαρμογής ή ότι θα πρέπει ο Ευρωπαϊκός Υπουργό Οικονομικών να αποφασίζει για το πώς θα δοθούν οι πόροι, όλα αυτά πρέπει να τα απορρίψουμε. Η αρχή της ευθύνη πρέπει να είναι η βάση της σκέψης μας και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέρμερ. Και τώρα η κυρία Θάβαλ, Γάρδια Θάβαλ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Από την αρχή της οικονομικής ε, κρίσης ε, έγιναν εμφανίσει οι αδυναμίες της αρχιτεκτονικής του ευρώ και ιδιαίτερω η ανάγκη να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε την ΟΝΕ. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι έγιναν βήματα προ αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στη μείωση των κινδύνων. Παρ' όλα αυτά, απομένει πολύ έργο να γίνει, να συμπληρώσουμε, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύηση Καταθέσεων ή, ε, ε, ή να διαθέτουμε πλέον ένα πραγματικό περιπολισμό τη ζώνη του ευρώ που θα επιτρέπει στι χώρε τη Ευρωζώνη να αντιμετωπίσουν καινούριε οικονομικέ κρίσει. Υπό την ομπρέλα τη ΟΝΕ, συζητούμε σήμερα την μεταρρύθμιση του ισχύοντο Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα ε, που ετέθησε λειτουργία το 2012 αλλά θα πρέπει να τροποποιηθεί. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός ε, θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωμή Τάξη. Αυτό θα επέτρεπε να τον διαχειριστούμε σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο. Και μεταξύ άλλων θα διευκόλυνε το συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και θα του έδινε μεγαλύτερη νομιμοποίηση και δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα ήταν ενδιαφέρον επίσης ο ευρωπαϊκός προπολογισμό να συνεισφέρει σε αυτό το μηχανισμό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έδινε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ασκεί δημοσιονομικό έλεγχο ε, και βέβαια να ελέγχεται από το ε, ε, ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς έχουμε καταγγείλει πολύ συχνά τις αυθαιρεσίες και τις υπερβολές που έγιναν υπό τις εντολές της Τρόικα. Ε, οι ζημιέ αναγνωρίστηκαν και από πολλούς ηθήνοντες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό στο μέλλον απαιτούμε τα ε, προγράμματα διάσωση ε, να λαμβάνουν υπόψη στο μέλλον και τι κοινωνικέ συνέπειε για να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Γνωρίζω ότι αυτά είναι συστάσει του Κοινοβουλίου βέβαια. Δεν έχουν νομική αξία. Έχουν όμως πολιτική αξία. Γι' αυτό το λόγο ελπίζω να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Λούκε. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην αρχή της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας υπήρξε παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθήκων για να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός. Σήμερα θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε με ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Άλλη μια παραβίαση των συνθήκων. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητε για τέτοια θέματα. Για να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό. Πουθενά σε ευρωπαϊκέ συνθήκε δεν λέγεται ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό. Άλλο ένα παράδειγμα ότι η Ένωση αφαιρεί τη μία μετά την άλλη από τι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Και τελικά όλα πάνε χειρότερα. Αν αναλάβει η Ένωση την ε, ευθύνη για την νομισματική πολιτική, ε, θα έχουμε άλλη μία κρίση σαν αυτή που είχαμε. Όταν, για παράδειγμα, πήρε η Ευρώπη την ε, ευθύνη για την πολιτική των προσφύγων, υπήρξε προσφυγική κρίση. Ποια αιτιολόγηση μπορεί να υπάρχει τώρα για να δώσουμε και για την μακροοικονομική σταθερότητα και για την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Αρμοδιότητε στην Ένωση είναι κατά του δικαίου, είναι κατά των συνθήκων. Δεν υπάρχει κανένα λόγο για να το κάνουμε. Αρμόδια και, ευρωπαϊκά, και με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκε είναι πάντα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Νίλ Στόρβαλτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ συχνά στην συζήτηση αυτή έχω την εντύπωση ότι έχουμε μια οικονομική αμνησία. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά την ιστορία και μιλάμε ως αν να εμφανίστηκαν αναντιστοιχίε και ανισορροπίε μόνο και μόνο με το ευρώ. Ας δούμε την Βρετανική ιστορία. 1956. Τι είχαμε τότε στη Βρετανία. Ένα έλλειμμα, καθώς επίσης και μια υπερτιμημένη λίρα και βέβαια μια οικονομική κρίση που ακολούθησε. Οι αναντιστοιχίε λοιπόν αυτέ, οι ανισορροπίε που έχουν προκαλέσει οικονομικέ κρίσει, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ίδια την ιστορία τη Ευρώπη. Και ένα Καλό γερμανό υπήρξε στην ιστορία αυτή, μόνο ότι επιτεθάμαστε πάρα πολύ στου Γερμανού, Ο Βίλι Μπραντ το 1969, ο οποίο σε μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε «Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 30% του πλεονάσματός μας στην Ευρώπη προκειμένου να αποτελέσει αυτό ένα πρώτο αρχικό κεφάλαιο για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο με όρο, είπε. Θα πρέπει εσεί να μπορείτε να διχειριστείτε από μόνοι σα τι οικονομίε σα. Και αν δεν είστε ικανοί για κάτι τέτοιο, τότε δεν θα πρέπει να έρχεστε εδώ πέρα και να ρίχνετε την ευθύνη σε άλλου για σφάλματα δικά σα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τα διδάγματα της ιστορίας και να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή είναι η κυρία Νιριάντα, 1,5 λεπτό. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Παρά το ότι δημιουργούμε άλλο ένα μηχανισμό και δεν έχει σημασία πώ τον αποκαλέσουμε, μηχανισμό σταθερότητα ή νομισματικό ταμείο, το ίδιο είναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει ανάγκη για ένα τέτοιο μηχανισμό, αλλά ω ε, Ιρλανδοί θα πρέπει να καταλάβετε γιατί θα ήμουν επιφυλακτικοί και όχι κατά ανάγκη υπέρ. Τι έγινε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, όπω και σε άλλε χώρε, όπω στην Ελλάδα, ακόμη πληρώνουμε για αυτήν την τρομερά απέσια διάσωση που ε, έγινε πριν από μερικά χρόνια και θα πληρώνουμε μέχρι το 2040. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να είμαστε τόσο αισιόδοξοι ότι ένα τέτοιο μηχανισμό θα λειτουργήσει προ το συμφέρον μα. Ιδιαίτερα αν δούμε το ότι πολλοί στην Ιρλανδία υποφέρουν ακόμη ε, από έλλειψη τη κατάλληλη κατοικία, δεν μπορούν να πάρουν ενυπόθηκο δάνειο από τι τράπεζε Έχουμε τα υψηλότερα επιτόκια για ενυπόθηκα δάνεια στον κόσμο. Έχουμε ε, πολλούς πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Δεν μπορούν να κερδίσουν τα προστοζήν. Γιατί λοιπόν νομίζουμε ότι θα λειτουργήσει ένας Πρέπει να είναι διαφανής, πρέπει να δράμε υπεύθυνο τρόπο. Και κάτι ακόμη που πρέπει να πω ιδιαίτερα για τις τράπεζες στη χώρα μου. Δεν πληρώνουν φόρο, δεκάρα, παρά το ότι βγάζουν ένα σωρό λεφτά πάλι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τα σπασμένα και τη λυπητερή. Γιατί πρέπει να είναι υπέρ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν νομίζω ούτε ότι οι Ιρλανδοί θα είναι ενθουσιασμένοι με αυτή την ιδέα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη, αλλά δεν νομίζω ότι ε, είναι καλά διαμορφωμένη πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Νιριάντα. Και ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Πεντιτσίνη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά πραγματικά σε τι χρησιμεύει ένα καινούριο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Μήπως πρέπει να διασώσουμε και άλλες γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε. Δώσαμε αρκετά ήδη. Είχαμε την φοβερή αυτή εμπειρία του 2010 με το πρόγραμμα διάσωσης, όπου με την δικαιολογία της διάθεσης Ισπανίας και της Ελλάδας 60 δισεκατομμύρια ευρώ χρειάστηκε να δώσουμε σε τρία χρόνια. Και καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα αυτά πήγανε κυρίω σε γαλλικέ και γερμανικέ τράπεζε. Ο γερμανικό και ο γαλλικό λαό ε, ούτε ένα ευρώ δεν είδε από τα χρήματα αυτά. Ένα τέτοιο νέο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ουσιαστικά θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στι ε, χώρε τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην ξεχνάμε πάλι ότι θα χρειαστούν και νέε χώρε να περάσουν από νέε μεταρρυθμίσει και νέε αναδιαρθρώσει που θα προκαλέσουν νέε πολιτικέ κρίσει. Και θα χρειαστεί να επιστρέψουμε εδώ πέρα για να ακούσουμε το μελλοντικό πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έρθει να μα ζητήσει συγγνώμη, όπω ζήτησε συγγνώμη ο Γιούνκερ από την Ελλάδα για τι καταστροφικέ συνέπειε που είχε εκεί η δράση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Είδαμε ότι ε, οι πολιτικέ λιτότητα αποτέλεσαν πραγματικά τροχοπέδι για την οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση και να έχουμε διευρυντικέ οικονομικέ πολιτικέ προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πραγματικά ζητήματα όπω η ανισότητα, η ανεργία και η έλλειψη οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πεντιτσίνη. Ο λόγος στην κυρία Έλισεν, τον κύριο Έλισεν. Μιλάμε για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα και τη μεταρρύθμιση του. Καθώ επίση και τη θέσπιση του Ευρωμοναδικό Νόμισμα, ενιαίο νόμισμα. Παλιότερα οι συνθήκε ήταν διαφορετικέ. Όταν εισήχθη το ευρώ έγινε μεγάλο λάθος. Δημιούργησε σημαντικά οικονομικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύξηση του χρέους και χαμηλή οικονομική ανάπτυξη. Χώρες εκτός του ευρώ, όπως η Νορβηγία και η Σουηδία, ε, υπέφεραν πολύ λιγότερο. Οι κάτω έχουν ε, δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ προς χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, ε, χώρες οι οποίες ε, δεν τήρουν τα κριτήρια σύγκλησης. Το ευρώ δεν είναι κάτι που μας δίνει χρήματα, μας κοστίζει. Το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεων. Και τα, Ευρωπαϊκά, και τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν θα έχουν πια δικαίωμα βέτο. Προφανώς είμαστε κατά. Προφανώς διαφωνούμε. Προτείνουμε ένα μηχανισμό σταθερότητας που θα ελέγχεται ε, από εθνικά κοινοβούλια μόνο. Ευχαριστώ. Can we fix it? Okay. Voimme Ωραία, συνεχίσουμε. Ο, ο κύριος Κάρας για δύο λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί εδώ και χρόνια να αναπτυχθεί περαιτέρω ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, διάσωση για να γίνει ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Το κάναμε στην έκθεση που κάναμε για τα αίτια και τι επιπτώσει τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση. Το κάναμε με την έκθεση πρωτοβουλία για τον έλεγχο της Τρόικα και το κάνουμε και σήμερα γιατί είμαστε πλήρως πεπισμένοι ότι πρέπει να εξαγάγουμε τα διδάγματα από την οικονομική κρίση και την κρίση του δημοσίου χρέους. Χρειαζόμαστε ισχυρότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση και θέλουμε και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση. Γι' αυτό τα θέλουμε όλα αυτά. Αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο όμως φυσικά πρέπει να βασιστεί στο ενωσιακό δίκαιο και να ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι απλώς να είναι διακυβερνητική πρωτοβουλία. Θέλουμε με αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο να βοηθήσουμε να υπάρχει σταθερότητα για τα κράτη-μέλη που θα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Αλλά αυτό θα γίνεται με ισχυρούς μηχανισμούς επιβολής μεταρρυθμίσεων και ε, καθηκόντων. Θέλουμε να έχει επαρκείς πόρους και να αποτελέσει υπορισμένες προποθέσεις και τμήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Να είναι μια ίστατη προσφυγή για να αντιμετωπιστούν, για παράδειγμα, ακόμη και προβλήματα της Τραπεζικής Ένωσης. Και αυτό θα κάνει πιο ανεξάρτητη και πιο σταθερή την Ευρώπη ούτως ώστε να ενισχύσουμε το ευρώ και ούτως ώστε χωρίς εξωτερική βοήθεια η Ευρώπη σε κατάσταση ανάγκης να μπορεί να παρέμβει και η Επιτροπή να βοηθηθεί στο έργο της για την εξυγίανση των καταστάσεων. Επιμένουμε και καλούμε τα κράτη-μέλη για να κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν επιτέλους το πλαίσιο για να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάρας. Και τώρα η κυρία Μπρέσο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, Προκαλεί γέλο όταν ακούμε εδώ πέρα τους εθνικιστικούς συναδέλφους οι οποίοι μιλάνε για την κυριαρχία των κρατών μελών ξεχνώντας βέβαια ότι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο το οποίο δεν πρόκειται να το ονομάσουμε και έτσι, γιατί ουσιαστικά θα εξακολουθεί να λέγεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός σταθερότητα. ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι στιγμή μέσω αποφάσεων που ελήφθησαν από τα ίδια τα κράτη-μέλη και όχι μέσω της συμμετοχής του μηχανισμού αυτού στην Ευρωπαϊκή Ενωμή Τάξη. Από αυτό ακριβώς, ε, από αυτή τη διαπίστωση ξεκινά η έκθεση αυτή, από τις δυσκολίες που προκλήθηκαν από την ε, διακυβερνητική διαχείριση του μηχανισμού αυτού και πρόθεση της έκθεσης είναι το νέο αυτό νομισματικό ταμείο να έχει την απαραίτητη νομιμοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε στα πλαίσια της έκθεσης αυτής ε, ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωμή Τάξη, μόλον ότι αυτό δεν γίνεται με απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο ακόμα από την έκθεση. Θα πρέπει να υπάρχει από το κοινό. Κοινοβούλιο επιτήρηση, εποπτεία, μεγαλύτερη λογοδοσία και από την, να ξεκινήσουμε και από την ίδια την ονομασία. Όπω είπαμε, δεν θα πρέπει να ονομαστεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αλλά θα πρέπει να εξακολουθεί να λέγεται Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση μέσω του μηχανισμού αυτού. Έχετε μία μπλε κάρτα, κυρία Μπρέσο. Τη δέχεστε? Από τον κύριο Έθεριτ. Από τον κύριο Έθεριτ, τη δέχεστε? Ναι, την έχετε. Ωραία. Είναι γνήσια ερώτηση. Χρησιμοποιήσετε μια λέξη που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είπατε ότι είμαστε υπέρ της ε, κυριαρχίας. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι είμαστε οπαδοί της κυριαρχίας. Είναι υποτιμητικός όρος. Είναι απλώς περιγραφικός. Γιατί μου έκανε εντύπωση. Ε, δεν είχα καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσω την μπλε κάρτα, αλλά πείτε μου τι σημαίνει η λέξη sovereignist, αυτός που είναι ο παδός της κυριαρχίας. Να απαντήσω Υπέρμαχος της εθνικής κυριαρχίας είναι αυτός που πιστεύει ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ανήκουν στα κράτη-μέλη ή να την χάνουν διαχείριση μόνο με τη διακυβερνητική μέθοδο. Όποιο είναι φεντεραλιστής όπως εγώ, πιστεύουμε ότι οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να περάσουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι θα πρέπει εκεί να την χάνουν διαχείριση. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με το νόμισμα. Äh, Ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε. Ο λόγος τον κύριο Κούσμιουκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα θα ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ. Ε, ο ισχύων διακυβερνητικό ε, μηχανισμός και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητα εξασφαλίζει ε, θα πρέπει να τεθεί σε κοινοτική βάση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Με αυτόν τον τρόπο ε, θα αυξηθεί η λογοδοσία. Ελπίζω ότι αυτό το Ταμείο και, άλλοι, και άλλες αλλαγές στην λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος ε, θα εφαρμοστούν και σε χώρες οι οποίες ε, ε, δεν βρίσκονται στην ε, Ευρωζώνη. Δεν θα πρέπει να μπλοκάρουμε την ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ζώνης του ευρώ, ούτε θα πρέπει να, μειωθούν ή να μειωθεί η δυνατότητα λήψη μειωθει η δυνατοτητα ληψης αποφασεων των χωρών που δεν βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ και για παράδειγμα η πρόσβασή τους σε, στα ταμεία και στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούσμιουκ. Ο κύριος Ομάρτζε έχει το λόγο. Merci. Πρόεδρε, η εμπειρία 10 ετών πολιτικών λιτότητας ε, κατέδειξε ότι είναι αναποτελεσματικές και αποτυχημένες σε όλη την Ευρώπη. Φαίνεται ότι δεν άρκεσε αυτή η εμπειρία. Ο Μακρόν και η Μέρκελ δεν βρήκαν τίποτα καλύτερο από το να ε, επινοήσουν ένα νέο αντιδημοκρατικό σύστημα θεσμό που είναι το Ευρωπαϊκό Νοσηματικό Ταμείο χωρίς κανένα έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα καταστρέψει όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα κράτη που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και θα λατήσει το κοινωνικό κράτος για να επιβάλλει ε, τις νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις. Στην πραγματικότητα ο Μακρόν και η Μέρκελ δημιουργούν ένα μηχανισμό που θα κατατρώει την δημοκρατία ε, και θα οδηγήσει αθλειότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Έθεριτς έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Όταν έχουμε δηλαδή χώρε, οργανισμού, επιχειρήσει και οικονομίε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε, εσεί μα λέτε ότι θα πάρετε τα χρήματα των φορολογουμένων και θα του τα δώσετε. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία κιόλα όταν ε, οι χώρε αυτέ εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη πάρα πολύ βοηθητικό εκ μέρου σα, πολύ εξυπηρετικό, αλλά οι χώρες αυτές, οι οργανισμοί, οι οικονομίες και επιχειρήσεις ε, αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες στα πλαίσια των περιορισμών της Ευρωζώνης, που εσείς τόσο και θελό τους εντάξατε στη ζώνη αυτή. Και αντί τώρα να έρθετε και να πείτε, πολύ ωραία τελικά το σύστημα δεν λειτουργεί, από ό,τι φαίνεται, οι οικονομίε αυτέ θα πρέπει να λειτουργήσουν αυτόνομα. Οι επιχειρήσει αυτέ, οι οποίε δεν είναι κερδοφόρε, θα πρέπει να καταρρεύσουν και να αντικατασταθούν από άλλε, γιατί ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο θα λειτουργούσε η ελεύθερη αγορά των κεφαλαίων. Αντί να λέτε αυτό το πράγμα, εσεί παίρνετε τεράστια χρήματα από του φορολογουμένου και προσπαθείτε να συντηρήσετε μια κατάσταση που δεν λειτουργεί από μόνη τη. και εγώ να σας δώσω, αν θέλετε, κάποιες συμβουλές για να σας βοηθήσω, αφού και εσεί το κάνετε. Θα σας πρότεινα, λοιπόν, το ακόλουθο να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε αυτό το, να επεμβαίνετε κατά αυτόν τον τρόπο στις αγορές. Δεν ποτέ δυνατόν να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο και να δαπανείτε δισεκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στους φορολογούμενους σε σχέδια τα οποία δεν λειτουργούν στην πράξη για μία ακόμα φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λεμπρετών, το αρχιτολόγο, για 1,5 λεπτό. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Ευρωζώνη είναι εγγενώς ε, ιδιαιτέρως εύθραυστη γιατί περιέχει πολύ ετερογενείς χώρες όπως η Γερμανία και η Ελλάδα για παράδειγμα το είπε το Νόμπελ Οικονομίας ο Αμερικανός Στίγλιτς και η επόμενη χρηματοοικονομική κρίση θα την ε, καταστρέψει από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί δίκτυα ασφαλείας όλο και πιο περιοριστικά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας δημιουργήθηκε το 2010 το 2013 έγινε Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και επειδή αυτός ε, θεωρείται ιδιαίτερα διακυβερνητικό, θέλουμε να τον μετατρέψουμε σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ακόμη πιο ενταγμένο. Αυτό το νέο μέσο θα είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό φορέα εντελώ. Άλλη μια επίθεση κατά τη εθνική κυριαρχία. Και γι' αυτό είμαι αντίθετο. Είναι προφανέ ότι αυτό ο μηχανισμό, όπω και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, θα δίνει βοήθεια στα κράτη-μέλη μόνο εάν κάνουν προγράμματα λιτότητας και ιδιωτικοποίησεων που θα τους επιβάλλει με βάση τα δόγματα της ε, άκρα της ε, νεοφιλελευθερίας τάσης. Δεν θα ήθελα του χρόνου και η Γαλλία να είναι παιχνιδάκι αυτού του μηχανισμού. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Στόλογιάν, δύο λεπτά. Βάρογκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευθύς εξ αρχής, να τονίσω ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει ένα χρηματοοικονομικό μέσο για να δίνει βοήθεια στα κράτη-μέλη όταν έχουν ανάγκη, η λογική λύση θα ήταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να περάσει από το διακυβερνητικό πλαίσιό του στην ενωσιακή ένωμη τάξη. Αυτό θα ήταν θετικό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και η έκθεση την οποία συζητάμε, υποστηρίζουν αυτή την ε, μετατροπή του μηχανισμού. Λυπάμαι όμως που το Συμβούλιο αποφάσισε να μην συζητηθεί η πρόταση της Επιτροπής. Στηρίζω την πρόταση της ε, Έκθεση ότι αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας να ε, μπορεί να χρηματοδοτήσει και κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη αλλά μόνο από την προπόθεση ότι θα υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα ούτω ώστε να ενταχθούν σε αυτήν. Ωστόσο αυτή η δυνατότητα πρέπει να δίδεται μόνο στα κράτη-μέλη που έχουν ήδη ε, λάβει την απόφαση να ενταχθούν στο ευρώ και που επίσης ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις και που εφαρμόζουν τα προγράμματα που έχουν αποφασιστεί από κοινού με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και υπάρχει και μια άλλη, έκθεση της, ε, μια άλλη πρόταση της έκθεσης που λέει ότι αυτός ο νέος μηχανισμός σταθερότητας θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα backstop, μια ίστατη καταφυγή δηλαδή. Και για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, ούτως ώστε έτσι να μπορούμε να εξηγιάνουμε καλύτερα το δεύτερο πυλώνα της ε, Τραπεζικής ε, Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λόγος στον κύριο Σίλβα Περέιρα. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να μεταρρυθμιστεί ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και να βοηθήσει ε, να γίνει πιο αποτελεσματικό ε, το ενιαίο ε, Ταμείο Εξυγίανση και να πραγματοποιηθεί η Τραπεζική Ένωση. Θέλουμε όμως ένα μηχανισμό σταθερότητας ε, πραγματικά ευρωπαϊκό, ενταγμένο στο ευρωπαϊκό δίκαιο και που να υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να είναι περισσότερο αυτόνομο σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συνεπώς να γυρίσει τη σελίδα των, της Τρόικα. Θέλουμε να κάνει περισσότερα για να στηρίξει τα κράτη-μέλη και να μάθει από τα διδάγματα των προγραμμάτων ε, ε, προσαρμογής του παρελθόντος. Δεν θέλουμε να... Ε, θέλουμε επίσης να κάνει μια σοβαρή αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων που συστήνει. Αυτά είναι τα μηνύματα της προσωρινής έκθεσης που θα εγκρίνουμε. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα έχουν ακούσει τη φωνή του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς έχει τώρα το λόγο. Για ένα λεπτό. Παρακαλώ, Grazie Κύριοι συνάδελφοι, πολλή μελάνη έχει χυθεί για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου στα χνάρια του μισητού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διέλυσε ολόκληρες χώρες και κοινωνίες με τελευταίο θύμα του το πειραματόζωον η ελλάς. αντί λοιπόν να αναζητάτε μηχανισμούς τύπου δελτα που φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό καλό θα είναι να χτυπηθούν οι αιτίες που οδήγησαν τις χώρες της ευρωζώνης στον κίνδυνο και στην πτώχευση. μία είναι η βασική αιτία και αυτή είναι η δομή αλλά και η πολιτική της ευρωζώνης ευρωζώνη που έχει δομηθεί για να εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντα ευρωζώνη η οποία λειτουργεί με βάση τον ζουρλομανδία του συμφώνου σταθερότητας που επιβάλλει λιτότητα και βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή. για το λόγο αυτό πρέπει να καταργηθεί το σύμφωνο σταθερότητας να μετατραπεί η ect σε ίστατο δανειστή να αποκεντρωθεί το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών και τα κράτη μέλη να ανακτήσουν την νομισματική τους κυριαρχία μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ect. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρωσάτη τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγγνώμη, την Επιτροπή μας για την προετοιμασία της έκθεσης αυτής, θεωρώ πραγματικά ότι σημειώνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδο αυτή τη στιγμή, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την οικονομική και νομισματική μας ένωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα αντικαταστήσει, θα απορροφήσει, αν θέλετε, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και θα αποτελέσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τη διαχείριση των κρίσεων. Η δράση αυτή ουσιαστικά έρχεται να καλύψει ένα πολύ σημαντικό κενό στο εφιστάμενο σύστημα διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Ποια καθήκοντα θα έχει ο μηχανισμό αυτό, Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ε, οικονομικέ δυσκολίε. Θα έλεγε κανεί ότι αυτό είναι ο ρόλο που ήδη επιτελεί το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, Σταθερότητα. Αλλά εγώ θα ήθελα να σα πω ότι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα επιτελέσει το καθήκον αυτό με έναν τρόπο πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Δεύτερον, θα αποτελέσει σίγουρα ένα μηχανισμό ασφαλεία για τι ε, τράπεζε που θα αντιμετωπίζουν ε, οικονομικέ δυσκολίε. Έτσι λοιπόν, χρηματοδοτώντα τα κράτη και τις τράπεζες θα καταφέρουμε τελικά να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο, αν θέλετε, το φαύλο θεσμό μεταξύ χρέους, οικονομικών κρίσεων και τραπεζών. Θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερος ο μηχανισμός αυτός. Δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει ένας μόνιμος μηχανισμός διαβίβασης πληρωμών. Και θα έχει και άλλα πλεονεκτήματα όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός ο μηχανισμός αυτός και αυτό διότι ανήκοντας επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, ο μηχανισμός λήψη αποφάσεων θα λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα και θα είναι σε θέση το νέο αυτό νομισματικό ταμείο να αντιμετωπίζει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο έγκαιρα τι οικονομικέ δυσκολίε και κρίσει στα κράτη-μέλη. Και κάτι ακόμα, δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο να θεωρούμε ότι θα έρθει να συναγωνιστεί το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει εδώ πέρα μία λύση έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε πρόσβαση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διεθνή οργανισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Τομά. Για ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η οικονομική κρίση του 2008 κατέδειξε τις επιπτώσεις, τις ε, καταστροφικές επιπτώσεις μιας ε, αντελούς ένωσης. Υπάρχει ελευθερία για τα κεφάλαια, αλλά αρνείται την οικονομική αλληλεγγύη. Οπότε η ολοκλήρωση της ΟΝΕ είναι αναγκαία και απαραίτητη για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη ε, οικονομική και νομισματική πολιτική. Ευχαριστώ του συνεισηγητέ για την εργασία του και χαιρετίζω το ότι το κείμενο αυτό εισάγει ένα δίκτυο ασφαλεία που επιτρέπει να παρέμβουμε με συντονισμένο τρόπο εάν υπάρξουν οικονομικέ κρίσει σε ένα κράτο μέλο, όχι μόνο προ όφελο του κράτου μέλου, για να αποφευχθούν οι αλυσιδωτέ αντιδράσει στην Ευρωζώνη. Όμω η δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου παραμένει στόχο υπό την ε, διακυβερνητική διαδικασία λόγω των κανόνων του, κοινό, του Συμφώνου Σταθερότητας και χωρίς να συμμετέχει στην διαχείρισή του ούτε να μπορεί να ελέγξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι συνέχιση των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόστηκαν κατά τη διαχείριση ιδιαίτερα της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Χωρίς διαφάνεια, χωρίς δημοκρατικό έλεγχο, η λογική ότι αυτό που πληρώνει θα αποφασίζει δεν θα είναι σωστή διακυβέρνηση τη νομισματική πολιτική. και θα έχουμε και πάλι τις ε, καταστροφικές επιπτώσεις αυτών των πολιτικών για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ε, παιδική φτώχεια. Ευχαριστώ. Τόμασιτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στην αρχή της έκθεσης λέγεται ότι η εισαγωγή του ευρώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται από το ποιο ρωτά. Α ρωτήσουμε του Ιταλού ή του Έλληνε. Το ευρώ έκανε ακόμη πιο συγκεντρωτική την Ευρωπαϊκή Ένωση και μείωσε τα περιθώρια ελιγμών για τα κράτη-μέλη. Το ίδιο θα επιτύχει ακόμη περαιτέρω αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα γίνει κάτι ακόμη ισχυρότερο. Κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται λογικό. Εάν υπάρχουν κρίσεις, πρέπει να είναι πιο ανθεκτική η Ένωση. Αλλά αυτή η πρωτοβουλία είναι μια απόπειρα οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων να γίνουν μόνιμοι και στην πραγματικότητα να ελέγχουμε τις λειτουργίες και το πώς δίνεται οικονομική βοήθεια. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Ποιετικά είναι. Δύο λεπτά. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου είναι λογική συνέπεια και λογική συνέχεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που δημιουργήθηκε μετά την, το ξέσπασμα της κρίσης του ευρώ. Όταν καταλάβαμε ότι πρέπει να διαθέτουμε ένα μηχανισμό σταθερότητας που να έχει δυνατότητα χρηματοδότησης εν το μέσο κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο αποτελεί τμήμα ενός ε, πιο μεγάλου παζλ και είναι σημαντικό, είναι σημαντικό στο μέλλον να λειτουργεί με τρόπο αυτόνομο και εντός του κοινοτικού κεκτημένου, όχι με τη μέθοδο της ε, διακυβερνητικής προσέγγισης. Οι αποφάσεις ε, θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση συγκεκριμένε αξίε και με βάση την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι από 27 ή 28 διαφορετικές ε, νομικές τάξεις. Υπάρχει περίπτωση τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν από μόνα τους με την ίδια αποτελεσματικότητα, τα ίδια κριτήρια και την ίδια αυστηρότητα. Για παράδειγμα, σε σχέση με την Γαλλία, τη Γερμανία και την Κύπρο. Θα είναι ισότιμη μεταχείρισή τους. Εμείς θέλουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να είναι αξιόπιστος και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα λειτουργήσει με ο τρόπο ομοιογενή, μακροπρόθεσμα και με βάση συγκεκριμένε αρχές και νόμους. Όχι με διαφορετικό τρόπο σε, σε ε, συνάρτηση με το ποια είναι η χώρα την οποία εξετάζει. είναι ένα πρόσθετο βήμα σε σχέση με την ε, Συμφωνία Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αναπτύσσει με αυτόν τον τρόπο την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του κύριο Γκάιερ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με εντυπωσιάζει η πολυγλωσία σας. Η πρόταση της ε, Κομισιόν να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός και να ενταχθεί στον ε, ενωσιακό, στην ενωσιακή ε, νόμη τάξη, ένομη τάξη είναι πολύ θετική γιατί έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε τον έλεγχο της λειτουργίας. Το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να αναβάλει περαιτέρω την εξέταση αυτού του θέματος. Είναι βασικό ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και χρειαζόμαστε ένα προπολογισμό της Ευρωζώνης με δυνατότητα σταθροποίηση όταν έχουμε συμμετρικές κρίσεις. Ο μηχανισμός αυτός είναι τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομιματικής τάξης. Δεν θα είναι κάτι που θα επικαλύπτει με τη λειτουργία του. Και πρέπει να έχει και τους αναγκαίους πόρους. Και γι' αυτό αυτή η ιδεολογική αιμονή για το 1% του ΑΕΠ, για τον ενωσιακό προπολογισμό που διάφορες ε, κυβερνήσεις ε, στηρίζουν στην διαπραγμάτευση για τις προοπτικές είναι λανθασμένη. Δεν θα πρέπει να είναι ταμπού η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να έχει δικής, δικούς του είδους πόρους ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε για παράδειγμα ένα φόρο επί των χρηματομισθωτικών ε, ε, συναλλαγών ή έναν ψηφιακό φόρο. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Κέλλη, δύο λεπτά. Παρακαλώ. Καλωσορίζω την εργασία για να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη ε, υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο να ε, ε, διαμορφώνουμε και εφαρμόζουμε τα προγράμματα οικονομική βοήθεια προ τα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Νομοσπονδιακό Ταμείο θα πρέπει να έχει περισσότερη ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων, αλλά το σημαντικό είναι η λήψη των αποφάσεων να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών. Ο επόμενο ενωσιακό προπολογισμό μπορεί να βοηθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσει πιο να προωθήσει την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων, να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των πολιτών μα. Νομίζω ότι το μέλλον τη ΟΝΕ θα είναι η ενίσχυση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να επανέλθει η εμπιστοσύνη του κοινού. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Επιπλέον, πρέπει να εστιάσουμε στην ανάπτυξη της ε, ε, Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Έχει τεράστιο δυναμικό να δημιουργήσει νέου μηχανισμού χρηματοδότηση των επιχειρήσεών μα και τη οικονομία μα και μπορεί να συμπληρώσει το πρόγραμμα επενδύσεων. Καλωσορίζω μια σειρά από διατάξεις του σχεδίου έκθεση, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να είναι δυνατή για όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για τα κράτη τη Ευρωζώνης. Καλωσορίζω επίση τι εκκλήσει που γίνονται ο μηχανισμό αυτό, να έχει επαρκή τεχνογνωσία για να έχει και το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης για να έχει τις σωστές διαδικασίες λήψη αποφάσεων. Καλωσορίζω την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου που προβάλλει θέση για το θέμα αυτό επειδή είναι ιδιαίτερα αργή η διαδικασία στο Συμβούλιο. Και πάλι, και όχι για πρώτη φορά, το Κοινοβούλιο επιδεικνύει πρωτοπορία προς το συμφέρον των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Σάντα. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόοδο για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου θα παραμείνει προβληματική, εκτό και αν ο πολιτικό διχασμός αυτή τη στιγμή, η πολιτική διχόνοια που παρατηρείται στη λήψη αποφάσεων επιληθεί. Θα πρέπει η Ευρωζώνη να βελτιωθεί και ουσιαστικά θα πρέπει να ενισχυθούν οι οργανισμοί εκείνοι που επιβλέπουν ε, την μακροοικονομική σταθερότητα και αποτρέπουν τι κρίσει. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερη λειτουργία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και ιδίω των μικρών και όχι μόνο για τις προτάσεις αυτές οι οποίες προχωρούν περισσότερο προς το φεντεραλισμό, πράγμα το οποίο δεν θέλουν ή θεωρούν ότι είναι αρκετά πρόωρο. Το να επιμένουμε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο ήδη από τώρα θα πρέπει να ενταχθεί στην κοινοτική μέθοδο ουσιαστικά τονώνει ακόμα περισσότερο τις αρνητικές στάσεις απέναντί του. Από την άλλη όμως Λέγεται ότι η διακυβερνητική μέθοδο θα επιβραδύνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Καλύτερα όμω να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο το οποίο θα λειτουργεί με βραδύτητα στην αρχή παρά ένα ε, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο το οποίο δεν θα είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σάιζενφελτ τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα που ε, εμφανίζεται είναι ότι ε, σε περιπτώσεις κρίσης ε, δεν υποφέρουν μόνο οι επιχειρήσει αλλά και οι πολίτες οι ίδιοι. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν ισχυρό μηχανισμό για να σταθεροποιεί τέτοιου είδου δημοσιονομικές διακοιμάνσεις. Επίσης, τα... οι λαοί χρειάζονται στήριξη σε, περιπτώσεις σε περιόδους ύφεσης. Ο μηχανισμός σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση σε αυτά τα προβλήματα. Ε, δεν θα σχολιάσω το θέμα του ονόματος γιατί υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα όπως για παράδειγμα η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η, η ομοφωνία θα έπρεπε οι ψηφοφορίε να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, όχι με ομοφωνία. Και τρίτον, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ποιο θα ήταν ο δικαιούχο τη ε, οικονομική στήριξη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Ο Ευρωπαϊκ... Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να διασφαλίζει ένα μηχανισμό προστασίας ε, για, τις... για περιπτώσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης. Ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να είναι μόνιμος επίσης και να συνδέεται στενά με την ίδια τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βάιντερη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεισηγητές και να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το ότι ε, ασχολούμεθα με ζητήματα τα οποία είναι πολιτικά ευαίσθητα. Το Συμβούλιο ούτε που έχει ξεκινήσει την εργασία για το ζήτημα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταρρυθμιστεί ο οργανισμό αυτό. Θα θέλουμε πραγματικά να έχουμε στο μέλλον εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε πιθανέ ε, οικονομικέ κρίσει. 19 μόνο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη της Ευρωζώνης. Άρα η οικονομική και νομισματική συνεργασία γίνεται δύσκολη σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης ή άλλων οικονομικών δυσχεριών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα μοντέλο συνεργασίας που θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη να βρίσκουν γρήγορε έγκαιρε λύσει σε περίπτωση δυσχεριών. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί πολύ καλή βάση για τη δημιουργία ενό τέτοιου μοντέλου. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και ως προς το όνομα το οποίο θα επιλέξουμε και αν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη όντως θα είναι ζωτική σημασία προκειμένου να ενισχύσει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε επικαλύψεις με άλλους σχετικούς οργανισμούς. Αν πραγματικά όμως τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν αποτελεσματικό και διαφανή μηχανισμό, τα όσα λέμε δεν αρκούν. Θα πρέπει να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες περισσότερο, να φύγουμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες εποπτείας, καθώς επίσης και λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Διευρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις αρμοδιότητες, θα πρέπει να πετύχουμε μια ισότητα ανάμεσα, μια ισορροπία μάλλον, ανάμεσα στην ανάληψη ευθύνης και τη λογοδοσία. Τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν περισσότερες ευθύνες απέναντι στου δικούς τους πολίτες και τους πολίτες άλλων κρατών μελών. Όταν μεταρρυθμίσουμε λοιπόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα, θα πρέπει να υποστηρίσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη βέβαια και όχι τι ε, τράπεζε. και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λογοδοσία που είδαμε στο παρελθόν. Α είμαστε, ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι στου πολίτε μα. Είδαμε ότι πολύ συχνά δίστανται οι απόψει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ενά λοιπόν μια χρυσή ευκαιρία να μεταρρυθμίσουμε τον υφιστάμενο μηχανισμό και να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητή σε. Ουδή θέλει το λόγο στο πλαίσιο, στα πλαίσια του Catch the Eye, δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ντομπρόφσκη, εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, άκουσα πολύ προσεκτικά τις παρεμβάσεις σας και η συζήτηση ήταν πραγματικά πολύ ζωντανή στηρίζουμε τους προβληματισμούς για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής ΣΟΝΕ στο μέλλον. Η δουλειά, ε, υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα. Η πρότασή μας για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο φαίνεται ότι είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση και να σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί αποτελεί ολοκλήρω, ε, ένταξη, μια ένταξη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου στη, στον κοινωτικό κεκτημένο θα βελτίωνε τις παρεμβάσεις του στο πλαίσιο της, ε, του συντονισμού των ε, δημοσιονομικών πολιτικών. Ε, το Συμβουλίο Κομισιών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Επίσης θα βελτιώσει την λογοδοσία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αυξήσει την δημοκρατική του νομιμοποίηση. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου δεν αφορούν μόνο τα κράτη-μέλη που είναι δικαιούχα, αλλά και συνολικά την ζώνη του ευρώ. Θα επιτρέψει επίσης βελτίωση της ε, διαφάνειας ε, ε, των δρασιών του. Η ένταξη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου στο κοινοτικό κεκτημένο θα αποτελεί και δείγμα της σημασίας που έχει λάβει η ζώνη του ευρώ τα τελευταία χρόνια. Τα κράτη-μέλη και το, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο προφανώς θα πρέπει να σέβονται τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι προφανές. Ευχαριστώ. Thank you very much, Vice President. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Μάνκα. Βλάντιμιρ, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω βέβαια και τον συνεισηγητή, τον Πέντρο Σίλβα Περέιρα, για την κοινή εργασία που κάναμε. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τους και οδησηγητές και όλους τους συνεργάτες μας για την εξαιρετική εργασία. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιλύσουν τους συστημικούς κινδύνους ευρωζώνης από μόνα τους. Δεν μιλάμε εδώ πέρα μόνο για πολυεθνικές, όπως είπε ο κύριος Μάρουσιτς. Αναφερόμαστε και σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίε θα μπορούσαν από οικονομική άποψη να ανθίσουν στα πλαίσια μια ευημερούσα οικονομία. Καταλαβαίνετε ότι ολόκληρε χώρε και περιφέρειε μπορούν πραγματικά να επηρεαστούν από την οικονομική κρίση που ξεκινάει από μια χώρα και απλώνεται σε άλλε. Χρειαζόμαστε μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε τέτοιε απειλέ. Ο υφιστάμενος διακυβερνητικός, η υφιστάμενη διακυβερνητική μέθοδος έδειξε τα όρια της όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων. Το να καταφέρουμε να εντάξουμε το μηχανισμό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη θα τον καταστήσει πιο αποτελεσματικό. Συνεπώς, θέλουμε να έχουμε μία αποτελεσματική βραχυπρόθεσμη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος, προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε τον μηχανισμό αυτό πιο φιλόδοξο για το μέλλον. Από μόνοι μα δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Μόνο από κοινού μπορούμε να προασπίσουμε πραγματικά την Ευρωζώνη και το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο, τον κύριο Μάνκα. Ολοκληρώνεται η συζήτηση στο σημείο αυτό. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την έκθεση του κυρίου Πιπέρα όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή μα, λοιπόν, τον κύριο Πίπερα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είμαστε μια Ευρώπη των ελευθεριών, των θεμελιωδών ε, αξιών. Είμαστε μια Ευρώπη που είναι υπέρ του θεμητού ανταγωνισμού, του ισότιμου ανταγωνισμού. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ισχυρή όταν δρά από κοινού. Οι αμερικανικοί δεσμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, οι δασμοί κατά των ε, χαλιβουργικών προϊόντων από πλευράς της Κίνας ε, δεν μπορούν να μας επηρεάσουν εάν, δράμ, δρούμε από κοινού. Φυσικά δρούμε με βάση τις εμπορικές ένωσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα τμήματα του κόσμου. Μια τέτοια βάση ακριβώς θέλουμε να διασφαλίσουμε με το νέο κανονισμό 868 σωστό ανταγωνισμό και στις εναέρες μεταφορές. Ένα τομέα όπου δεν ισχύουν μέχρι στιγμής οι κανόνες του ΠΟΕ. Περί τίνο πρόκειται. Σε άλλα τμήματα του κόσμου οι αεροπορικές ε, εταιρείες επιδοτούνται με μεγάλα ποσά. Τόσο πολύ που στρεβλώνεται ο ανταγωνισμό.